Bien, mesdames, messieurs, αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Έχουμε βέβαια μισή ώρα καθυστέρηση. Δεν μπορούμε να ε, προχωρήσουμε μετά τις 7. Ε, πρέπει να σταματήσουμε στις 7 η ώρα. Άρα θα πρέπει να μειώσουμε τον ε, χρόνο της συνεδρίασης Πρώτα απ' όλα θα συζητήσουμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και κατόπιν για τους ενδεχόμενου νέους ίδιους πόρους του ενωσιακού προϋπολογισμού. Οπότε, καλό όσους θα πάρουν το λόγο να είναι σύντομοι. Καταρχάς να σας χαιρετήσω ολόθερμα ε, να χαιρετήσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα θέλω να χαιρετήσω την κυρία Ευγένια Αγγέλοβα, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της ε, Εθνοσυνέλευσης της ε, Βουλγαρικής Δημοκρατίας. Θα προεδρεύσει το δεύτερο γύρο της συζήτησης. Είναι πολύ σημαντική η συνάντησή μας για να σφυριλατηθούν οι δεσμοί μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα για δημοσιονομικά και φορολογικά θέματα. Η πρώτη συζήτησή μας αυτή τη Διακοινοβουλευτική Επιτροπή θα ασχοληθεί με το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Πρέπει να ανταποκριθούμε στι ε, αναδυόμενε προκλήσει και στι νέε προτεραιότητε και στη χρηματοδότησή τους. Είναι λοιπόν ε, στιγμή κλειδί για να ακουστεί η φωνή των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να εκπονήσει δύο στρατηγικέ εκθέσει πρωτοβουλία. Μία για το πολιτέ πλαίσιο και δεύτερον για την ε, μεταρρύθμιση των ίδιων πόρων. Οι δύο αυτέ ε, εκθέσει θα εγκριθούν στι επιτροπέ αυτή τη βδομάδα και το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Και ε, θυμίζω ότι οι δασμοί ε, μειώνονται συνέχεια και δεν είναι παρά 10% των πόρων του προπολογισμού. Θέλουμε να παρουσιάσουμε λοιπόν τις απόψεις του Κοινοβουλίου πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώσει την πρότασή της, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί τον ε, προσεχή Μάιο. Λοιπόν, μερικά θέματα διαδικαστικά τώρα. Πρώτα απ' όλα πώς θα παίρνετε το λόγο υπογραμμίζω ότι όπως συνήθως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να δώσουμε το λόγο σε όσο δυνατόν περισσότερους ε, συμμετέχοντες ακόμη και αν έχουμε περιορισμένο χρόνο διότι όπως ξέρετε η Ολομέλεια κράτησε περισσότερο επειδή έχουμε πολλούς συμμετέχοντες δεν θα είναι δυνατόν να λάβουν όλοι το λόγο σήμερα αλλά θα υπάρξει δυνατότητα αύριο το απόγευμα να λάβουν και άλλοι το λόγο. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Δύο λεπτά αγαπητοί συνάδελφοι. Θα σας αναφέρετε ο χρόνος, θα βλέπετε το ρολόι. Όπως ε, πάει η συζήτηση θα δούμε αν θα χρειαστούν περαιτέρω περιορισμοί στο χρόνο ομιλίας. Και θα είμαστε πολύ αυστηροί με το χρόνο ομιλίας. Είμαστε υποχρεωμένοι. Πάνω στα γραφεία σας έχετε δύο κάρτες. Μία πράσινη με αυτή μπορείτε να ζητάτε το λόγο για την πρώτη συζήτηση. Η δεύτερη είναι κίτρινη για τους νέους ίδιους πόρους. Εάν θέλετε να παρέμβετε, παρακαλώ να ε, συμπληρώσετε τις κάρτες και να τη δώσετε στους κλητήρες. Αυτό ισχύει και για τους εθνικούς και για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσουμε ο χρόνος ομιλίας να είναι ως εξής. Δύο εθνικοί βουλευτές και κατόπιν ένας ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Αν χρειαστεί, κυρία Πρόεδρε, ίσως χρειαστεί να... Εάν χρειαστεί, ίσως προσαρμόσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, ξεκινώντας να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές για την έκθεση πρωτοβουλίας για τις πολιετές προοπτικές και πρώτα στην κυρία Ιζαμπέλ Τομά. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από εδώ, δηλαδή ως Ευρωβουλευτές, θεωρούμε ότι είστε το ίμιση των προσπαθειών μας. Πραγματικά πρέπει να αλληλοσυμπληρώνουμε τις προσπάθειές μας. Γιατί εσείς ε, ψηφίζετε τις δαπάνες και εμείς ψηφίζουμε Συγγνώμη, εσείς ψηφίζετε τα έσοδα και εμεί ψηφίζουμε τις δαπάνες. Πρέπει λοιπόν να συνεργαζόμεθα. Αλλά πολύ σπάνια έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να ανταλλάξουμε απόψεις. Πρέπει να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία, αυτή η σύμπνοια. Γιατί ορισμένοι θα ήθελα να πιστέψουμε ότι είμαστε αντίπαλοι. Συχνά και απόλυτα αντίπαλοι. Όμως αυτό δεν ισχύει. Όπως έχει τώρα ο ενωσιακός προϋπολογισμός, ίσως να έχετε την εντύπωση όταν αυξάνετε τους εθνικούς προϋπολογισμούς ότι μειώνεται τον ενωσιακό και εμείς έχουμε την αντίστροφη εντύπωση ότι όταν αυξάνουμε τον ενωσιακό μειώνουμε τους εθνικούς. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί αυτή η παρεξήγηση. Δεν θα μιλήσω εγώ για τους ίδιους πόρου. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό για μα. Πρέπει να αλλάξει η δομή των εσόδων του ενωσιακού προπολογισμού. Των εσόδων της Ένωσης γενικότερα. Και γι' αυτό ως Επιτροπή Προπολογισμών προτείναμε το θέμα του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου να εξαρτάται από τη βελτίωση και την τροποποίηση της δομής των εσόδων της Ένωσης. Κάποιοι μπορεί να λένε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν ισχύουν. Δεν το κάνουμε επειδή θέλουμε να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρω ο προπολογισμό τη Ένωση. Στόχο μα είναι να διασωθεί ο ενωσιακό προπολογισμό. Και μέσω τη διασώσεω του θα σώσουμε και την ίδια την Ένωση. Γιατί αυτά που κάνουμε τώρα, όλα αυτά που ακούμε, όχι ίσω όλα, όχι. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20 κατώτερο του προηγουμένου αν λάβουμε υπόψη την ένταξη της Κροατίας το παρόν πλαίσιο λοιπόν δεν τα βγάζει πέρα γιατί υπάρχουν τόσο πολλές περικοπές και διάφορα που προκύπτουν στην πορεία που έχουν επιπτώσεις. Και τελικά τις υφίστανται οι συμπολίτε μας που θα έπρεπε να είναι οι κύριοι δικαιούχοι της Ένωσης. Υπάρχει το πρόβλημα των περικοπών στην ε, πολιτική συνοχή, ε, στην πολιτική έρευνα, στους φοιτητές ε, που θέλουν να λάβουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Έρασμος και άλλους. Αλλά κυρίως υπάρχουν προβλήματα με το προσεχές πολιτές πλαίσιο αλλά και με το υπάρχον. Αυτό που εκτελείται τώρα εμπεριέχει τρομερές αντιφάσεις. Και ακούνε οι συμπολίτε μας και πολύ αντιφατικά επιχειρήματα και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Από τη μία τους αναγγέλουμε ότι πέρα από τις παραδοσιακές πολιτικές της Ένωσης, γεωργία, συνοχή κτλ. Η Ευρώπη θέλει να ασχοληθεί και με πολλά άλλα θέματα. Θα ασχοληθεί με τους πρόσφυγες, με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με την άμυνα, ιδιαίτερα με, την, με τον κλάδο της παραγωγής ε, αμυντικών εξοπλισμών και τέτοια, με πολλά άλλα θέματα. Βεβαίως, όλοι θέλουν να ασχοληθεί και με στο μίση η Ένωση, χωρίς να αυξηθεί και χωρίς να τίθεται το θέμα αύξησης από αυτούς που κάνουν τέτοιες διακηρύξεις του προπολογισμού. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε σοβαροί, και θέλουμε ως Επιτροπή Προπολογισμών να είμαστε, τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βεβαίω συμφωνούμε ότι δημιουργήθηκε το Σέγγεν χωρίς να θέσουμε το θέμα των συνόρων. Σε ένα διεθνές πλαίσιο δυσχερές, σίγουρα χρειαζόμαστε να επενδύσουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα. Αλλά, παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς επιπλέον πόρους. Χωρίς φράγκο παραπάνω. Γι' αυτό θέτουμε το θέμα με σοβαρό τρόπο ενός ευρωπαϊκού προπολογισμού που να είναι στο ύψο των διακηρυγμένων φιλοδοξιών. Τώρα, στη συζήτηση με το Συμβούλιο. Πολλά κράτη-μέλη αναγγέλουν ότι το κενό των 12 δις που θα προκύψει από την, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρειάζεται να καλυφθεί μέσω αύξηση των εσόδων. Μας είπαν ότι θα πρέπει απλώς να αποφασίσουμε ποιες προτεραιότητες θα διατηρηθούν και ποιες περικοπές. Περικοπές σε μερικά από τα παραδοσιακά στηρίγματα της Ένωσης. Προειδοποιώ. Η Επιτροπή Προπολογισμών δεν ενέκρινε ακόμη την έκθεση, οπότε όλα όσα σας λέω είναι σε υποθετικό λόγο, γιατί θα ψηφίσουμε την Παρασκευή στην Επιτροπή και το Μάιο στην Ολομέλεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα υπάρξει ευρεία συνένεση. Αυτό αναμένουμε. Οι παραδοσιακές λοιπόν πολιτικές της Ένωσης που είναι πολιτικές αλληλεγγύης όπως η συνοχή, το κοινωνικό ταμείο, η γεωργική ε, πολιτική. Όλες αυτές είναι πολιτικές που συνδέονται με την ε, ενιαία αγορά. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι έχει έννοια εάν θέλουμε να έχουμε μια φιλόδοξη προοπτική για την Ευρώπη να κάνουμε περικοπές ε, στα ίδια τα θεμέλια της Ένωσης και του προπολογισμού της. Για να αυξήσουμε γενικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μα δεν θα μπορέσει να γίνει μεγαλύτερο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα υπονομεύοντας τα θεμέλια του. Τουλάχιστον εμείς έτσι νομίζουμε. Όπω σας είπα, αυτές οι πολιτικές είναι η έκφραση της κοινοτική αλληλεγγύη. Σχετίζονται με την ε, ενιαία αγορά. Είναι πολιτικές τι οποίες υπολογίζουν οι συμπολίτε μα και είναι και πολιτικές επενδύσεων, ιδιαίτερα η πολιτική συνοχής. Είναι η κυριότερα πηγή επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ψιθυρίζουν ότι μία λύση θα μπορούσε να ήταν η πολιτική συνοχής να περιοριστεί στις πιο μειονευτικές περιοχές αλλά μακροπρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα, ίσως όχι βράχη πρόθεσμα, το αποτέλεσμα αυτό μια τέτοια πολιτικής θα είναι ότι τα κράτη-μέλη που δεν θα υποφελούνται από αυτήν την πολιτική να μην θέλουν πλέον να τη χρηματοδοτήσουν και να κυριαρχήσει η λογική του καθαρού εισφορέα. Θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις είναι επεπαλαιωμένες. Όλοι ωφελούμεθα από τις επενδύσεις αυτές που γίνονται, όπου και αν γίνονται. Όλοι είτε είναι καθαροί συνεισφορείς, είτε καθαρά ωφελούμενοι. Δέκα λεπτά δεν είπατε. Α, καλά. Α, με συγχωρείτε. Καλά, λοιπόν, καταλήγω. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε. Καταλήγω λέγοντας ότι Κάναμε έναν απλό υπολογισμό. Η διατήρηση χωρίς αυξήσει των υπαρχουσών χρηματοδοτήσεων στις παραδοσιακές πολιτικές, κάτι που ήδη θα δημιουργήσει χέρε αν υπάρξουν αυξήσει συν οι πολιτικές που, αυξ... που εισήχθησαν εκ των υστέρων και που είναι χρήσιμε. όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της ανεργία των νέων η χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες ή η χρηματοδότηση για τα σύνορα. Και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαιτήσει του Συμβουλίου για τις μελλοντικές πολιτικές άμυνας, του κλάδου της άμυνας, καταλήξαμε σε έναν απλό υπολογισμό για το, πολιετές, για το επόμενο πολιετές πλαίσιο θα πρέπει να φτάσουμε στο 1,3 στο όριο του 1,3 του ΑΕΠ, με ιδιαίτερα δηλαδή συγκρατημένη προσέγγιση. Δεν ξέρω, ίσως κάποιους να σας ε, σκανδαλίσει, γιατί ορισμένοι θεωρούν δεν πρέπει να υπερβούμε το 1%, αλλά σας ε, διαβεβαιώνω ότι είναι ιδιαίτερα μετροπαθής αυτή η εκτίμηση, αλλιώς θα πρέπει να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι αυτή η γνώμη της πλειοψηφίας των Ευρωβουλευτών. Ο κύριος Γιάνν Ολμπρεχτς είναι για 7,5 λεπτά τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες ε, συμπληρωματικές παρατηρήσεις από πλευράς μου. Σας συνεισηγητής μαζί με την κυρία Τωμά. Ε, είμαι μεν Πολωνός, θα μιλήσω όμως αγγλικά για να διευκολύνω την όλη συζήτηση. Ποιο είναι το πραγματικό ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε τι θα συμβεί επακριβώς μετά το 2020, αυτό είναι το ερώτημα. Τι θα συμβεί μετά το 2020 με τον ενωσιακό προπολογισμό και τις διάφορες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Και φυσικά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι αρνητική. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει και με τους Βρετανούς μετά το Μάρτιο του 2019 και η όλη συζήτηση που σας την περιέγραψε η κυρία Τομά αφορά το τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020. Αυτό είναι το πρώτο. Τι περιμένουμε. Πώς περιμένουμε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020. Και τι θα θέλαμε να κάνουμε μαζί και ποιες θα είναι οι κοινέ δράσεις και βέβαια πόσο θα κοστίσουν όλες αυτές. Υπάρχει αρκετό χρήμα για να τα κάνουμε όλα. Όχι βέβαια. Άρα είναι και θέμα πολιτικών αποφάσεων και μετά το 2020 θα μπορούμε να καλύψουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα, διαρθρωτικά ταμεία. Θα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. 1η Ιανουαρίου του 2021. Για να είμαστε έτοιμοι θα πρέπει να τα έχουμε ολοκληρώσει όλα το αργότερο στα μέσα του 2019. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε τουλάχιστον ο κανονισμός για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να έχει περατωθεί πριν από τις ευρωεκλογές αν δεν έχει περατωθεί σχετική εργασία, θα χρειαστεί χρόνος, θα χρειαστεί ίσως και το 2019 και το 2020, οπότε θα έχουμε καθυστερήσει. Δεν είναι κάτι βέβαια καινοφανές αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα θέλαμε να το αποφύγουμε και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αμέσω μετά το 2020. Αυτά λοιπόν είναι τα πολιτικά ζητήματα. Και το ερώτημα είναι, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε γρήγορα, μέσα σε 6-7 μήνες ενώ συνήθως η διαδικασία αυτή ε, απαιτεί δύο χρόνια. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, διότι θα απαιτήσει συμφωνία μεταξύ κυβερνήσεων, κυβερνήσεων των κρατών μελών δηλαδή, αλλά και τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με τον ετήσιο προϋπολογισμό η ψηφοφορία γίνεται με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Η διαδικασία είναι διαφορετική. Μετά το Συμβούλιο, εφόσον έχει αποφασίσει με ομοφωνία, θα στείλει το σχέδιο προπολογισμού στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα μπορεί να πει ναι ή όχι. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε φυσικά, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε τώρα και να μην περιμένουμε το Συμβούλιο. Ήδη από τώρα είμαστε εμεί έτοιμοι, όμω θέλουμε και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια να δείξουν ότι διαθέτουν πολιτική βούληση και θέλουν να ε, είναι και αυτοί έτοιμοι το στομότερο δυνατόν. Διότι αν δεν προχωρήσουμε όλοι μαζί δεν θα είμαστε έτοιμοι πριν τις ευρωεκλογέ. Όταν λέω εμείς ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι έτοιμη πριν την αλλαγή σκητάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν την αλλαγή Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα είμαστε έτοιμοι. Άρα πολιτικά μιλώντας, τα πάντα θα είναι ανοιχτά ή θα ξανανοίξουν. Θέλουμε λοιπόν να τα έχουμε ολοκληρώσει. Θα τα συζητήσουμε και αύριο τα περί του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Η συζήτηση για το πολιετέ αφορά όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική συζήτηση, η οποία αφορά το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit. Και δεν θα μα απασχολήσει μόνο το κόστο, αλλά και το τι θέλουμε να κάνουμε μετά το Brexit από κοινού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Όλμπριχτ. Τώρα το λόγο έχει ο εισηγητή για τον προπολογισμό του 2019, ο κ. Ντανίλα Βιώτη, είχε 10 λεπτά στη διάθεσή του, δέχτηκε να περιοριστεί ο χρόνο του στα 7 λεπτά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι Ιταλό. θα ξεκινήσω λοιπόν την ομιλία μου στα Ιταλικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Αρτουή, θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφους που είναι εδώ παρόντε σε αυτήν ε, την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική ε, Εβδομάδα που πάντοτε ήταν σημαντική γιατί μας βοηθάει να καθορίσουμε κοινέ γραμμές ε, στο έργο μας. Όπως είδατε, είπαν και οι δύο συνεισηγητές, κύριε Τωμά και ο κύριος Σόλπιχτ, πολύ ξεκάθαρα ότι είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε φέτος για το πολιτισμικό πλαίσιο και πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Το 2018 είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη χρονιά επομένω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει τη διαδικασία για το πολιτές νοσονομικό πλαίσιο και εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε παράλληλα και τις διαπραγματεύσεις για το Brexit. Ο προπολογισμό του 2019 τώρα είναι μια διαδικασία που μας φέρνει αντιμέτωπους με πολλές προκλήσεις για το κοινοβουλίο μας είναι η τελευταία δυνατότητα που έχουμε για να παγιωθεί αυτή η συνέχεια των προτεραιοτήτων μας. Και εγώ θα εστιάσω σε τρεις πολιτικές προτεραιότητες πέραν των παραδοσιακών δράσεων που ήδη περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο προπολογισμό, έρευνα, ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων έχουμε όμως τρεις βασικές προτεραιότητες. Πυλώνας Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δικαιωμάτων το πρώτο. Μέσω των πολιτικών αυτών, των κοινωνικών πολιτικών, μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Εξού και είναι σημαντική αυτή η προτεραιότητα. Επίσης, διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Ενώ παράλληλα πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε τις ε, χώρες ε, προέλευσης, από τις οποίες φεύγουν οι μετανάστες δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια, τη ρίζα του προβλήματος της μετανάστευσης και βέβαια θα πρέπει να ενισχύσουμε και την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Γκέτεμπορκ αποφάσισαν να ενισχύσουν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Πέρυσι είχαμε εξαιρετική εργασία του κ. Μούρεσαν, του συναδέλφου μας, που οδήγησε σε αύξηση του σχετικού προπολογισμού, κάτι που θα συνεχιστεί και φέτος με την ε, εγγύηση για την νεολαία. Αυτή ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερη προτεραιότητα, τρίτη ε, γραμμή, τρίτο κονδύλι του προπολογισμού. Δεν καλύπτεται με επαρκείς πιστώσεις δυστυχώς. Θα πρέπει τον ΝΕΑΖΟ, τη Frontex ε, και το Ταμείο για την Ένταξη των Προσφύγων να ενισχυθούν σε ό,τι διαφορά την τρίτη προτεραιότητα, την αμυντική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια προπαρασκευαστική ενέργεια 12 εκατομμύρων ευρώ. Ε, η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη, οι Υπουργοί Άμυνας ε, έχουν προσυπογράψει τη σχετική αυτή πρωτοβουλία. Πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε πρόοδο και στο μέτωπο της άμυνας. Στόχος είναι να είμαστε πρωταγωνιστές ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Κατάλληλα προσαρμοσμένα τα εργαλεία και τα μέσα ε, στις ε, φιλοδοξίες και τους στόχους μας. Γι' αυτό απαιτείται ένας στέρος προπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Άρα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Δεν αρκεί η δίκαιη επιστροφή. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έχουμε και κάποια εξωτερικά χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν υπόκειται όμως στο δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλουμε να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση. Αν και κάποιες φορές τεχνικώς αυτό είναι αναγκαίο, όπως είδαμε κατά το παρελθόν όταν χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Το θέμα είναι πάντως να ιεραρχήσουμε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και να προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε με την ανάλογη πρικοδότηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανισορροπία σε ό,τι αφορά αυτά τα μέσα τα συμπληρωματικά. Εκεί κλείνει η πλάστικα περισσότερο. Τελικά έχουμε μια τεχνοκρατική Ευρώπη πολύ απομακρυσμένη από τους πολίτες. πολλές φορές δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις πιέσεις του Συμβουλίου. Και πολλά ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετώπιση την ανεπάρκεια των κρατών μελών, χωρίς όμως να δίνονται συμπληρωματικοί πόροι. Εσείς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς από τα εθνικά κοινοβούλια, θα πρέπει να δρέψετε τους καρπούς ε, των έργων των προηγούμενων ετών και των ημερίδων που συναντιόμαστε εδώ. Και όταν επιστρέψετε στις πρωτεύουσέ σας θα πρέπει να ασκήσετε πιέσεις στις κυβερνήσεις σας, ώστε όλοι, όλες οι κυβερνήσεις και η δική μου, ανεξαρτήτως του τι πρόσωπο θα έχει μετά τις εκλογές του Μαρτίου, ώστε όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις να προσπαθήσουν να βγουν από το σημερινό αδιέξοδο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό. Ελπίζω η συζήτηση που θα ακολουθήσει να μας δώσει τη δυνατότητα να χαράξουμε μια στρατηγική ε, κοινό έργο. Ξέρετε ότι είμαστε οι άμεση εκπρόσωποι των πολιτών μετά τις ευρωεκλογές ή τις εθνικές εκλογές και αυτό που επιθυμούμε είναι να έχουμε έναν προπολογισμό που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Ευρώπης για να επικρατήσει κάποια ηρεμία στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βιώτη που μίλησε για τις ε, επιπτώσεις ε, της αυστηρότητας ό,τι αφορά το πολιτικό πλαίσιο. Εφόσον ε, έχουμε εντάξει σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο τις ε, δαπάνες της επταετίας και συνεχώς υπάρχουν ε, απρόβλεπτες καταστάσεις που ανακύπτουν. Έχουμε εδώ πέρα, βλέπετε και το σχεδιάγραμμα, το λεγόμενο δημοσιονομικό γαλαξία με τις διάφορες ε, δομές που λειτουργούν παράλληλα και δεν ξέρω αν τα εθνικά κοινοβούλια διατηρούν ε, τον έλεγχο, γιατί έχουμε αρκετά χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, δεν ξέρω κατά πόσο και εσείς έχετε τον έλεγχο αυτών των μέσων, πάντως σας σίγουρα δεν τον έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να επιστρέψουμε στην δημοσιονομική ενότητα. Ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Βιώτη για την παρέμβασή σας. Τηρήσατε και το χρονικό όριο. Ο Γιώργη Ολέ έχει το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Θα μιλήσω αγγλικά. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσω τους ε, συναδέλφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και θέλω να επισημάνω ορισμένα στοιχεία που αφορούν ε, το ερχόμενο ΠΔΠ και που είναι σημαντικά για την πολιτική μας ομάδα. Πρώτον, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 περισσότερο από κάθε άλλο τέτοιο δημοσιονομικό πλαίσιο προπολογισμό ε, θέτει τις βάσεις ε, για την επόμενη επταετία και αφορά κυρίως ε, το πολιτικό όραμα. Ο προπολογισμό μεταφράζει λοιπόν ε, ε, τις πολιτικές προτεραιότητες και το όραμα που έχουμε σε οικονομικά στοιχεία. Πρέπει λοιπόν πρώτα να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, τι δεν θέλουμε πλέον να κάνουμε και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού θέλουμε να κατευθυνθούμε σε πολιτικό επίπεδο, ποιοι είναι οι πολιτικοί μας στόχοι και πώς θα τους μεταφράσουμε σε αριθμητικά στοιχεία. Το βασικό μέλημα είναι να έχουμε κοινού στόχους και να αποφασίσουμε πώς θα χρηματοδοτηθούν. Το ερώτημα είναι όμως, υπάρχουν αυτοί οι κοινοί στόχοι. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κοινό όραμα για τη μορφή που θέλουμε να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα χρόνια. Έχουμε κάνει μία σε βάθος συζήτηση για το όραμά μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν περάσουμε στη, σε βάθος συζήτηση για το πολιτές δημοσιογραφικό πλαίσιο και τελικά καταλήξαμε σε κοινά συμπεράσματα. Παρόλε τι καλέ προθέσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ διατηρώ τι αμφιβολίε μου. Δεύτερον, για να γνωρίζουμε που κατευθυνόμαστε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο ενωσιακό προπολογισμό ανέρχεται στο μόλι 1% του κοινού ακαθάριστου ε, εισοδήματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα έχουμε και αρνητικές ε, τάσεις τα τελευταία χρόνια, παρότι ε, συνεχώς ανακύπτουν νέες προκλήσεις και αυτό το φαινόμενο έχει ενταθεί. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, δεν υπάρχουν υψηλά επίπεδα φιλοδοξία στον τρέχοντα προπολογισμό, ούτε ε, προσήλωση προ ε, μια πιο ισχυρή και ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θεωρώ ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να επιδείξουμε φιλοδοξία και να προτείνουμε έναν ε, κατάλληλο, κατάλληλο επίπεδο πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση που να δείχνει μεγαλύτερη προσήλωση και φιλοδοξία σε ό,τι αφορά μια πιο ισχυρή και ολοκληρωμένη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, κατά τη γνώμη μας, ο προβλησμός πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ε, ορίζεται με ένα πολύ οπλωρωμένο και σφαιρικό τρόπο. Ο νοσικός προβληματισμός, λοιπόν θα πρέπει να ε, προβλέπει και μια ευρωπαϊκή ανταπόκριση ε, και ανάληψη δράση σε ό,τι αφορά τον ε, στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί πραγματικά είναι ε, πιεστικές αυτές οι προκλήσεις. Προτείνουμε λοιπόν το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να εστιάσει την προσοχή του σε ε, στόχους όπως ε, η καταπολέμηση της αύξηση ε, των ανισοτήτων μεταξύ κοινοτήτων και επικρατιών εντό Ευρωπαϊκή Ένωσης, ο προπολογισμό να επικεντρώνεται στην προστασία του πλανήτη, με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης. Όπως ξέρετε, με τη Συμφωνία των Παρισίων έχουμε υπογράψει και κυρώσει την ε, Συμφωνία των Παρισίων. Όμως τώρα πρέπει να γίνουν όλα αυτά πράξη. Πριν από μερικά χρόνια, ο κ. Βαρόσο πρότεινε τουλάχιστον 20% ε, των δαπανών αφορούν ε, το κλίμα. Τώρα αυτό θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, να γίνει τουλάχιστον 30% στο επόμενο ΠΔΠ. Προκειμένου να λάβουμε υπόψη τις νέες ε, διεθνείς ε, δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ε, προανέφερα, τη Συμφωνία των Παρισίων και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και θεωρούμε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού των κλιματικών δαπανών θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να διευκρινιστεί. Για να λαμβάνει όλες τις διαστάσεις υπόψη, και για να διασφαλίσετε και σωστή παρακολούθηση της εφαρμογής του. Μια άλλη προτεραιότητα θα είναι να επενδύσουμε περισσότερο στο μέλλον μας, στις μελλοντικές γενναίες, μέσω προγραμμάτων και δράσεων όπως το πρόγραμμα Έρασμος ή το πρόγραμμα απασχόλησης ε, της νεολαίας, ε, να επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνολογία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων για τις μελλοντικέ υποδομές και επειδή αμελούμε κάποιες φορές τον πολιτισμό, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον πολιτισμό. Δαπάνες για την έρευνα και καινοτομία θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, με ιδιαίτερη έμφαση ε, στις ε, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές. Μόλις το 9% των συνολικών δαπανών έρευνας και καινοτομίας αφορούν ε, την πράσινη έρευνα και ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Ε, επίπεδα αντίστοιχα με αυτό του προηγούμενου προγράμματος. Και για την ε, διευκόλυνση σύνδετο στην Ευρώπη και εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο ε, στην διασυνορική διάσταση, τα πράσινα ενεργειακά και μεταφορικά δίκτυα. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο σημαντικό τομέα είναι η μετανάστευση και η κοινωνική ένταξη. Και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί όταν εξετάζουμε το θέμα τη μετανάστευση, κυρίω επικεντρωνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ε, ασφάλεια των συνόρων και στην σφράγισή τους. Όμως θα πρέπει ε, να εξετάσουμε και την ευφυή διαχείριση των συνόρων προκειμένου ε, να διασφαλίζεται και η νόμιμη και ασφαλής ε, διέλευση, να έχουμε κατάλληλα προγράμματα επανακατάστασης ή εναλλακτικά συστήματα για να υποδεχόμαστε ε, τους ε, πρόσφυγες και κοινωνικές πολιτικές που θα βοηθούν τους μετανάστες και τους ε, πρόσφυγες να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας. Και κάτι τελευταίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και οικονομικά και πολιτικά να παρουσιάζει συνέπεια και συνοχή. Τα όσα λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε Εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τα προβάλλουμε και προ τα έξω, εκτό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατία, ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά βιώσιμη ανάπτυξη. Και για να τα κάνουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν ισχυρότερο τέτοιο φορέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σολέ. Και τώρα να δώσω το λόγο σε εσάς συναδελφοί, σε όσους έχουν ζητήσει. Πράσινα, πράσινες κάρτες πήρα μόνο από εθνικούς βουλευτές και γερουσιαστές. Η συνάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής... Α, βλέπω μερικές πράσινες κάρτες. Πρώτα απ' όλα η κυρία ε, Αν Μιλντερ από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά ο πυρήνας του προπολογισμού είναι η επιλογή. Αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν να κάνουν με τα ζητήματα του προπολογισμού. Πάντα στην πολιτική αυτό είναι δύσκολο να κάνει κάποιο επιλογέ και στο Κοινοβούλιο έχουμε και αυτή την αρχή ε, ότι όταν κάποιο προτείνει που θέλει να δαπανίσει χρήματα πρέπει να προτείνει και από πού θα γίνουν οι περικοπές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι γενικά πρέπει να ε, δαπανούμε περισσότερα και πρέπει να πείσουμε και τι κυβερνήσει μα ότι αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά αν θέλετε να δαπανίσετε περισσότερα, αυτό σημαίνει ότι τα εθνικά κοινοβούλια είτε θα πρέπει να κάνουν τα ίδια περικοπέ ή να επιβάλλουν νέου φόρου. Και κανεί δεν γίνεται δημοφιλή όταν κάνει τέτοιε προτάσει. Γιατί θα πρέπει να κάνουμε περικοπέ ε, στην υγεία ή να αυξήσουμε του φόρου. Δεν γίνεται έτσι δημοφιλή η Ευρωπαϊκή κανουμε περικοπε στην υγεια η να αυξησουμε του φορου δεν γινεται ετσι δημοφιλη ευρωπαικη ενωση έχουμε και μια μικρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λόγω του Brexit. Αυτό λογική συνέπεια είναι και προέκταση να γίνει και μικρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προπολογισμό τη. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει αυτό. Φαντάζομαι ότι το Μάιο θα γίνουν νέε προτάσει για νέε δαπάνε, αλλά θα σα ε, συνιστούσα πρώτα να εξετάσετε την αποτελεσματικότητα ε, των ε, σημερινών δαπανών. Συχνά βλέπουμε φωτογραφίε άδειων λιμένων, αερολιμένων, σκορπισμένα ευρωπαϊκά χρήματα, ευρωπαϊκοί πόροι. Ούτε έτσι γίνεται δημοφιλή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για του φόρου και του ίδιου πόρου θα έλεγα να μην ξεκινήσετε από εκεί γιατί ο Ολλανδός αν ακούσει ότι έρχονται ευρωπαϊκοί φόροι θα φύγει τρέχοντας. Καλό είναι λοιπόν να μην ακολουθήσετε αυτήν την άκουσα. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Ευρώπη. Πρέπει να λύσει τα μεγάλα διασυνοριακά προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους ε, τα κράτη-μέλη. Κλίμα, ασφάλεια, μετανάστευση. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθείτε σε ό,τι αφορά τον επόμενο προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Mulder. Μαργαρίδα Μαρκές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους προηγούμενους ε, ομιλητές, εισηγητές και σκιώδεις για, που μας μίλησαν για την προετοιμασία του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Να αναφέρω πρώτα την συνοχή. Συμφωνώ με τις ανησυχίες της ε, Ιζαμπέλ Τομά. Θα αποδυναμώσουμε την πολιτική συνοχής. Όχι, πρέπει να είναι ισχυρή. Πρέπει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια νέα γενιά πολιτικών συνοχής, όπου θα ενταχθούν και άλλες στην πολιτική συνοχής. Για παράδειγμα, η ένταξη των μεταναστών, όπως είπε ο Ισπανός συνάδελφος, στις μεγάλες πόλεις, για να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση. Αυτά είναι εγχειρήματα συνοχής αυτές της μεγάλου πόλεις. Πρέπει λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και όχι να αποδυναμωθεί η πολιτική συνοχής. Δεύτερον, ήδη οι πόροι. πρέπει να δώσουν περισσότερα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν προτάσεις. Και πρέπει να αρχίσει μια διαπραγμάτευση για να θέσουμε τα κράτη-μέλη ενώπιον των ευθυνών τους. Αυτά που δεν θέλουν να δώσουν περισσότερα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πρέπει να τα πείσουμε ότι έχουμε αυτές τις νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα, άμυνα και προστασία των συνόρων. Αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν όλες τις χώρες και αυτές που δεν θέλουν να δώσουν παραπάνω. Ο Πρωθυπουργό μας τόνισε ότι είναι ανοιχτός επί της επιβολής φορολόγησης επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και για την οικονομία του άνθρακα. Για τους ίδιους πόρους, κυρία μου, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Καλώς, λέει η κυρία Μαρκές. Επίσης, το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο δημιούργησε μια ειδική επιτροπή για να παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές πλαίσιο πλαίσιο. Είτε τώρα που καθορίζεται το πλαίσιο, το γενικότερο, είτε κατόπιν για τη διαπραγμάτευση μεταξύ Πορτογαλίας και Ένωσης. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος ε, ε, Χωσέ Μανουέλ Φερναντές που είναι Πορτογάλος Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ. Όλοι ξέρουμε ότι είμαστε διατρεφιλόδοξοι στην Ένωση. Και η στρατηγική 2020 είναι η απόδειξη, η οποία στρατηγική πέρασε ε, με μεγάλη συνένεση. Την ενέκριναν όλα τα κράτη-μέλη, όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Με 1% του ΑΕΠ προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα. Μα δεν ανταποκρίνεται στους στόχους, στις φιλοδοξίες. Αλλά ξέρετε, άβολη τη βρίσκω αυτή τη συζήτηση. Δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Δεν θα έπρεπε να γίνεται ε, με αφαιρέσεις, αλλά από κάτω προς τα πάνω. Κάθε κράτος μέλος να πει τι θέλει. Και βεβαίως μετά να συμφωνήσουμε. Για την έρευνα, για παράδειγμα, και την καινοτομία. Για τους νέους. Για τη συνοχή. Για τους μετανάστες την αλληλεγγύη και μετά να κάνουμε την πρόσθεση πόσο κάνει τούζο, πόσο κάνει το άλλο και να δούμε που καταλήγει. Αλλά αντίθετα, ξεκινάμε το 1%, άντε 1,1 και το κοινοβούλιο λέει όχι 1,3. Για πολύ απλούς λόγους. Γιατί οι στόχοι της στρατηγικής 2020 δεν έχουν εφαρμοστεί και αντιμετωπίζουμε και νέες προκλήσεις. Ε, μετανάστευση, ασφάλεια, άμυνα. Αν θέλουμε να είμαστε στο ύψος των προσδοκιών των συμπολιτών μας, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και όλα αυτά. Και κατόπιν θα έχουμε και την τρύπα 10 δις από τον Brexit. Και δεν είναι και τόσο πολλά το 1,3, είναι 175 δις. Ετησίως. Δεν είναι τόσο τερατώδες, αλλά θα μας επιτρέψει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ναι, κατά λίγο, κατά λίγο. Και γιατί να είναι κατά του Συμβουλίου, κατά το Συμβούλιο σε αυτά. Αν δούμε τις διακηρύξεις όλων, μα όλων των κρατών μελών, δεν θα έφτανε ούτε το 1,3 για ε, τις προσδοκίες που δημιουργούν στους ε, συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βαζίλ Κοκός από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για το δημοσιονομικό μέλλον της Ένωσης ε, δεν μπορεί να γίνει σωστά αν δεν έχουμε αντλήσει διδάγματα από την τρέχουσα περίοδο 2014-2020 και το τρέχον πολιετές, όπου τα κοντήλια ε, που δόθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις και να καλυφθούν οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, επειδή είναι χαμηλό το επίπεδο των διαθέσιμων κονδυλίων, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις της Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν μεταρρύθμιση της δομής των ευρωπαϊκών εσόδων, όπως την προτείνει και η ομάδα των πυρονομόνων υπό τον Μάριο Μόντι το 2016 για να μπορούμε να έχουμε ένα πιο σταθερό, προβλέψιμο, βιώσιμο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να να έχουμε ένα πραγματικό σύστημα ίδιων πόρων, πραγματικών ίδιων πόρων, που θα είναι ένα μεγαλύτερο κομμάτι του ενωσιακού προϋπολογισμού. Τουλάχιστον το μισό σε σχέση με τις ε, εθνικές συνεισφορές. πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα δεν δείχνουν να εμπιστεύονται και τόσο πολύ τις ε, πολιτικές που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό διότι τα τελευταία χρόνια είχαμε κάποιους μηχανισμούς χρηματοδότηση, κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία που προσπαθούν να καλύψουν ένα τεράστιο φάσμα στόχων. Δεν υπήρχε όμως και απαραίτητη ευθύνη. Θα πρέπει με διαφανή τρόπο να εξηγήσουμε στους πολίτες και να κάνουμε πιο λιανό αυτό το σύστημα το τόσο πολύπλοκο. Θα πρέπει να έχουμε έναν προϋπολογισμό που θα είναι πιο κοντά στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Επόμενος ομιλητής, ο Λεοπρόεδρος Ζωέλ Ζήκο, Γενικός συζητητή για τον Προϋπολογισμό από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος ε, για το ίδιους αλλά έχουμε καταλάβει όλοι πόσο θα περιπλέξει τα πράγματα από χώρες του Ενωμένου Βασιλείου. Είναι όμως και μια ευκαιρία για να ξανασυζητήσουμε κάποια ζητήματα. Και θα ήθελα να επιμείνω, το έκανα και περισσότερο για τις εκπτώσεις αυτές τις ε, επιστροφές. ένα δισεκατομμύριο παραπάνω πληρώνουμε ε, σε σχέση με άλλες μεγάλες χώρες όπως ε, η Γερμανία και έχουμε και το ΦΠΑ. Επίσης μια ειδική μορφή έκπτωσης. Ε, εμείς θέλουμε να αυξήσουμε ως Γαλλία τη συνεισφορά μας, όμως αυτό θα είναι υπό και χαίρομαι που στη συμφωνία μεταξύ ε, σοσιαλδημοκρατών και χριστιανοδημοκρατών ε, στη Γερμανία φαίνεται επίσης να υπάρχει βούληση για αύξηση της ε, γερμανικής συνεισφοράς. Θέλω να είμαι σύντομος, υπήρξαν πολλά που αναφέρθηκαν σημαντικά και στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Θα πρέπει όμως ε, και οι πιο πλούσιοι να βοηθήσουν την ανάπτυξη των πιο ε, φτωχών. Αυτό είναι η ίδια η πεμπτουσία της αρχής της αλληλεγγύης. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε λοιπόν να επανακατευθύνουμε τους διαφορετικούς πόρους περισσότερο προς, τους, ε, προς τα μέρη και να αποπλήττονται από την παγκοσμιοποίηση αυτή που έχουν επιλέξει να κάνουν πολιτικές διαρθρωτικές, μακροπεριφερειακές στρατηγικές για παράδειγμα που προωθούν την ολοκλήρωση. Είναι κάποιες πίστες αυτές που σας αναφέρω. Ευχαριστώ. Κύριε Ντέρ Γκαρθιαθάμπαλ, έχει τώρα το λόγο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για προπολογισμό και για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλέ φορέ λέμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερο. Εμένα. Ε, Πάντοτε μου προκαλεί την προσοχή αυτή η φράση. Πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Αυτό είναι αυταπάτη, είναι φενάκι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη είναι αυτό πρέπει είναι σαφέ του. Και το έρετημα είναι, αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερα χρήματα στον ενωσιακό προπολογισμό. Αλλιώ θα πρέπει να δεχθούμε ότι θα πρέπει να γίνουν λιγότερα από πλευρά πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα υπάρχουν επαρκή πόροι. Και η απόδειξη ότι αυτό που λέω ισχύει είναι το ε, πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο το τρέχον. Αντιμετωπίσαμε την κρίση τη μεταναστευτική και την προσφυγική. Χρειάστηκε να φτιάξουμε ένα σχέδιο επενδύσεων, να δημιουργήσουμε ε, το σώμα αλληλεγγύη. Τι χρειάστηκε να γίνει. Ε, έπρεπε να πάρουμε χρήματα από άλλα προγράμματα και να περιοκόψουμε προπολογισμού άλλων προγραμμάτων. Άρα δεν γίνεται να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Και πρέπει γι' αυτό να ληφθεί μια απόφαση και οι βασικές αποφάσεις ε, έχουν ως γνώμονα. Θέλουμε να έχουμε και γεωργική πολιτική στο μέλλον. Θέλουμε να τη διατηρήσουμε ε, στο επίπεδο το ευρωπαϊκό ή θέλουμε να την επανακρατικοποιήσουμε. Επίση, άλλο θέμα. Θέλουμε να έχουμε μια περιφερειακή πολιτική ε, συνοχή ή θα αποφασίσουμε ότι ένα μέρο τη Ευρώπη δεν θα αποφελείται πλέον από την πολιτική συνοχή, διότι τελικά πράγματι είναι το θέμα ε, να υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των πιο πλούσιων και των πιο φτωχών. Αλλά πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Δεν θα πρέπει λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στερήσουμε την πολιτική συνοχή. Το ίδιο ισχύει και με την Επιτροπή Άμυνα, την Επιτροπή Έρευνα και Ανάπτυξη. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πολλά παραδείγματα αναφέρθηκαν. Δεύτερο, σχόλιο που θέλω να κάνω, δεν έχω και πολύ χρόνο. Αευελιξία. Διότι θα πρέπει να αποφασίσουμε τώρα τι θα γίνει τα επόμενα δέκα χρόνια. Και επειδή δεν έχουμε όλε τι απαντήσει, γιατί ούτε και τι ερωτήσει δεν τι έχουμε ακόμα, γι' αυτό χρειάζεται ευελιξία. Και τελευταίο σχόλιο. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν τι ευρωεκλογέ του 2019. Και είναι σημαντικό που είναι εδώ τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί πρέπει να ασκήσουν οι εθνικοί βουλευτέ πιέσει ε, στι κυβερνήσει του. Η Πορτογαλία με την Επιτροπή Ελέγχου των διαπραγματεύσεων ήταν κάτι σημαντικό ε, και πρέπει το παράδειγμα τη Πορτογαλία να το ακολουθήσουν και άλλοι. Μην χάσουμε δύο χρόνια για να υιοθετήσουμε τι πολιτικέ που χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζον Λάχαρτ έχει το λόγο τώρα από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και την Αρμόδια Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα ορισμένε παρατηρήσει. Ε, βλέπω ότι το σημείο εστίαση στι Βρυξέλλε επικεντρώνεται κυρίω ε, στο Brexit και κατά βάση στον αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως θα πρέπει συνεχώς ε, να τονίζουμε, όπως έγινε και στην αποστολή ε, στο Δουβλίνο, ότι θα πρέπει να αναδείξουμε και τις προεκτάσεις του Brexit στην Ιρλανδία που σίγουρα θα επηρεαστεί όπως και άλλες χώρες από τον Brexit. Ανάλογα με τον τύπο του Brexit και τη μορφή που θα πάρει αυτό το Brexit, θα επηρεαστεί αντίστοιχα και ε, η οικονομία μας που τώρα ανακάμπτει. Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι μεταξύ 4 έως 9% ετησίως. Από τη στιγμή που θα γίνει το Brexit μέχρι το 2030. Οπότε δεν είναι μόνο ο αντίκτυπος στον ενωσιακό προπολογισμό ή στον Ιρλανδικό προπολογισμό, αλλά και σε συγκεκριμένε περιφέρειες, γιατί στην Ιρλανδία ο αντίκτυπο θα είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα κάτι ακόμα για του πυλώνε και τι προτεραιότητε που αναφέρατε. Σαφώ και η μετανάστευση ε, είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα ορισμένα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη ε, γραμμή. Μιλήσατε για την άμυνα για τις στρατιωτικά ουδέτερες ε, χώρες, ακόμα και ο όρος άμυνα έχει ε, πολιτικό πρόσημο, όμως ε, ξέρω ότι είναι σημαντική επένδυση και στην κυβερνοασφάλεια αντίστοιχα, οπότε και διατύπωση είναι σημαντική κατά την λήψη και παρουσίαση αποφάσεων επί του προπολογισμού. Να μην μιλούμε δηλαδή μόνο για τον στρατιωτικό αμυντικό εξοπλισμό, να εντάσσουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια και την κυβερνοασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Δελμάρ Αλγούλο, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Χαίρετε. Το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι τμήμα του οράματός μας, μιας πιο ισχυρής και πιο ενοποιημένης Ευρώπης και μια πιο ισχυρή και ενωπημένη Ευρώπη θα είναι περισσότερο σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Ο ενωσιακός προπολογισμό πάντα τα περασμένα χρόνια μπόρεσε να ε, βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη και την ενιαία αγορά. Αυτός είναι ο κεντρικός του στόχος. Και θέλουμε αυτός ο ρόλος να διατηρηθεί και στο μέλλον γιατί μια ενιαία εσωτερική αγορά είναι το κύριο ε, προτέρημά μας για να υπάρξει ευημερία και της Ευρώπης και των ε, πολιτών της. Θεωρούμε λοιπόν ότι κάτι που είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την ενιαία αγορά είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ε, η βιώσιμη ανάπτυξη και πολύ συγκεκριμένα για την Ισπανία η κοινή γεωργική πολιτική και οι δαπάνες συνοχής. Αυτές οι δαπάνες όμως είναι και πηγή πόρων στην ουσία. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια κατεδείχθη η σημασία της πολιτικής συνοχής και της γεωργικής πολιτικής. Αυτές ήταν οι κύριες πηγές επενδύσεων στην Ένωση. Στήριξαν την σύγκληση διαφόρων περιφερειών που βράδυ πορούσαν αλλά βοήθησαν και ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Άρα στην ουσία δημιούργησαν πόρους. Οπότε οι πολιτικές αυτές πρέπει να είναι ένα όργανο περισσότερης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, αλλά και ως πηγή πόρων. Είναι μια επένδυση ουσιώδης στο μέλλον της Ευρώπης, στο μέλλον της ευημερίας των συμπολιτών μας. Τώρα, για το νέο σύστημα ίδιων πόρων. Έχει ε, γίνει πολύ περίπλοκη αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Το πολιετές πλαίσιο μετά το 2020 είναι μια καλή ευκαιρία για την απλούστευση των εσόδων του ενωσιακού προπολογισμού να σταματήσουν οι επιστροφές και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να βασίζεται στο ΑΕΠ. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο πιο συγκεκριμένος δείκτης που θα χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Brexit δεν είναι λόγος ε, να κόψουμε τις ε, σχέσεις μεταξύ μας. Ε, μπορούμε να το αδράξουμε, να δράξουμε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ακριβώς ε, τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενοχίσουμε προτεραιότητες και μετά να βρούμε τους κατάλληλους πόρους ε, για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ε, με βάση και τις εθνικές συνεισφορές και τους ιδίους πόρους. Όμως θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε αυτό το όραμα. Κάποιες φορές νιώθουμε ότι έχουμε την αντίστροφη κατάσταση. Πρώτα να έχουμε τα χρήματα και μετά να δούμε ποιος έχει το πάνω χέρι προκειμένου, προκειμένου να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα, το οποίο έχει συμβεί πολλές φορές ε, ε, σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά το παρελθόν, το έχετε δει. Όμως ε, το MFF ε, πρέπει ε, να συνδυάζει τους στόχους και τους πόρους. Πρέπει να εξηγούμε με τον κατάλληλο τρόπο τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε για να έχουμε και την νομιμοποίηση της κοινή γνώμης. Δεν γίνεται να έχουμε προκαταβάλει τις τις προτεραιότητες για να ε, βρούμε και τους αντίστοιχους στόχους. Η αρχή της ε, ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει και αυτή να γίνει σεβαστή. Όμως το βασικό είναι να μείνει ζωντανή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρή. Γιατί υπάρχουν σαφείς ε, λαϊκιστικές και ευρωσκεπτικιστικές τάσεις και έτσι το σύστημα θα πρέπει να λειτουργήσει υπέρ και όχι κατά της Ένωσης. Βασική στόχη του προπολογισμού, ε, η τόνωση και χρηματοδότηση της συνοχής, μακροοικονομική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενίσχυση ε, του μηχανισμού ανακατανομής ή αναδιανομής για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες και το πλέον βασικό η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών και υπηρεσιών, μάλλον ενίσχυση των ευρωπαϊκών προϊόντων, Ευχαριστώ. Merci. Je vais demander à Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο τώρα στους δύο εισηγητές. Δυστυχώ ε, δεν έχετε πολύ χρόνο στη θέση σας. Δύο λεπτά έκαστο, αν είναι δυνατόν. Θέλετε να απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Όπως ε, ήρθεστε στην πολιτική, δίσταται οι απόψεις και γι' αυτό είναι και τόσο πλούσια, πλούσιος ο πολιτικός βίος. Ε, μπορούμε να σας πούμε τι θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε περισσότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε μεγαλύτερο προπολογισμό. Όμως, πολύ ξεκάθαρα μπορούμε να πούμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε όχι τον ίδιο προπολογισμό, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο σε σχέση με πριν από το Brexit. Ή θέλετε μετά το Brexit να αλλάξει το επίπεδο εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών. Αν θέλετε να μείνουμε λοιπόν στα ίδια επίπεδα, είναι απολύτως απαραίτητο να προσδιορίσουμε το κοστολόγιο και να βρούμε τους πόρους, είτε από τις εθνικές εισφορές, είτε με ιδίους πόρους. Το θέμα δεν είναι να έχουμε μεγαλύτερο προπολογισμό, δεν έχουμε τέτοια φιλοδοξία. Θέλουμε όμως ως κοινοβούλιο και από όλες τις πολιτικές ομάδες, έτσι, θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν οι κυβερνήσεις αποφασίσουν και έχουν αποφασίσει να προσθέσουν νέα στοιχεία όπως η άμυνα, η ασφάλεια, εμείς τίθουμε το εξής ερώτημα. Εντάξει, να συμφωνήσουμε. Αλλά εφόσον υπάρχουν νέες προκλήσεις, δεν πρέπει και αυτές να καλυφθούν από χρηματοδότηση. Όταν προσθέτουμε πολιτικές και νέες προκλήσεις, πρέπει να προσθέσουμε και πόρους. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να διευκρινίσουμε τους στόχους και ε, τη χρηματοδότηση με έναν εύλογο τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Τωμά. Για ένα λεπτό. Μάλιστα, για ένα λεπτό. Να διευκρινίσω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό. Θέλουμε να τον αφήσουμε περίπου στα σημερινά του επίπεδα. Πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί όχι μόνο δεν είμαστε ετεθειμένοι να μειώσουμε το επίπεδο φιλοδεξιών μας, και δεν το λέω εγώ αυτό, και το Συμβούλιο το λέει. Αλλά επιπροσθέτως προτείνονται νέες ε, προκλήσεις και τομείς ε, υπευθυνότητας ευθύνης μάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω ακριβώς αυτό. Ότι δεν πρόκειται για... Δεν μπορούμε να έχουμε νέα προγράμματα, νέους ε, τομεί ευθύνης χωρίς νέους πόρους. Και κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και εγώ και ο Γιάνν Όλμπρικτ και όλα τα μέλη ε, της Επιτροπής Προπολογισμών είναι απολύτως ειδηθημένα να έρθουν σε επαφή μαζί σας όλη αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε ε, στο δεύτερο τμήμα της σημερινής συνεδρίασης, να, κάνουμε, να απευθύνω μια έκκληση. Είστε μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και μιλούμε για την προσταθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχουν προκλήσεις που αυτή τη στιγμή εν και της παγκοσμιοποίησης ε, δαπανώνται σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο και δεν ε, καλύπτουν όλες τις δυνατότητες τους. Μήπως θα έχει έρθει η ώρα να δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να το πω με άλλα λόγια, αν αυξηθεί ε, ο ευρωπαϊκός προπολογισμός αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη πτώση των εθνικών προπολογισμών. Αυτό ε, μας επιτρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Σε κάποιους ε, τομείς ίσως διάστημα, μετανάστευση, Οπότε εκεί απαιτείται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε μία μεταφορά πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δείξουμε ότι σφαιρικά η αύξηση των δημοσίων δαπανών ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενωσιακού προπολογισμού δεν οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων δαπανών στην Ευρώπη. Κλείνω την παρένθεση, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Alors, nous, nous devons changer les, les rapporteurs. Έχουμε τώρα νέους εισηγητές. Λεβαντόφσκι και Ντεπρέ παρακαλώ να έρθουν στο Προεδρείο. Ο κύριος Διώτη φεύγει. Και θα έρθει ο κύριος Λαμασού. Thank you, Honorable Chair. Um, Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά η δυνατότητα να συμπροεδρεύσω μαζί με τον κύριο Αχτσουή τη συνεδρίαση αυτή ε, των ε, Επιτροπών Προπολογισμού των Εθνικών Κοινοβουλίου με την Επιτροπή Προπολογισμών της Ένωσης. Ξέρετε ότι έχουμε αναλάβει την Προεδρία για πρώτη φορά ως Βουλγαρία. Παρά το ότι είναι λοιπόν η πρώτη μας Προεδρία, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται. Τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καταδείξει επανειλημμένα ότι δεν ε, θεωρούν ε, αυτού και αλλήλου ως αντιπάλους. Μπορούμε να συνεργαστούμε προ το κοινό συμφέρον των συμπολιτών μα. να ενισχύσουμε τη δημοκρατική του φωνή. Οι κοινέ μα προσπάθειε, μπορεί να είναι ένα ισχυρό όργανο για να προσεγγίσουν οι πολίτε στην Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, η ενίσχυση αυτής της ε, επικοδημητικής συνεργασίας θα πρέπει να είναι ορόσημο και παράδειγμα για όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Φυσικά η εργασία των ε, Ευρωπαίων κοινοβουλευτικών είναι πολύ σημαντική τώρα που υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός και λαϊκισμός. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου πώς όρισε ο Ζακ Ντελόρ το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνεργασία ανταγωνισμός που ενισχύει και αλληλεγγύη που ενώνει. Πρέπει να βρούμε πώς θα συνεργαστούμε για να βρίσκουμε τις βέλτιστες λύσεις που να αντανακλούν την κοινή βούληση όλων των Ευρωπαίων που επιθυμούν να προχωρήσουμε υπερβαίνοντας τις δυσχέρειες. Οι νέες γενιές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να παίξουν ε, σημαντικό ρόλο δίδοντας νέα ενέργεια και νέες ιδέες για τη μεταρρύθμιση της Ένωσης για να ανταποκριθεί πλήρως στις υψηλές προσδοκίες των συμπολιτών μας. Ανησυχητικό ιδιαίτερα είναι ότι για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Οι νέοι ενήλικες μπορεί να είναι φτωχότεροι από τους γονείς τους. Σήμερα πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Ένωση είναι είτε ιδιαίτερα απόμακρη ή ότι παρεμβαίνει ιδιαίτερα στην καθημερινότητά τους. Θέλουν η Ένωση να δώσει συγκεκριμένες λύσεις ε, στην κρίση που αντιμετωπίζουμε, είτε είναι οικονομική, κοινωνική, είτε πολιτιστική. Το πιο σημαντικό θέλουν απαντήσεις για το πώς θα βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο η Ένωση και αναμένουν σαφείς απαντήσεις. Άρα σε εμά απόκειται, σε εμά όλους τους κοινοβουλευτικούς να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις και να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς στις απαντήσεις αυτές. Αλλιώς θα είμαστε στο επίπεδο το, το μετα, της μετα-αλήθειας. Χρειάζεται λοιπόν αλληλεγγύη και ελευθερία, αλλά επίσης ευημερία και βιωσιμότητα. Να θυμόμαστε τις αρχές που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους και τις κοινέ επιτυχίες μας. Σε αυτή τη συγκυρία η Ένωση χρειάζεται ισχύ και αποφασιστικότητα για να διατηρηθεί η ενότητά μας και να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Στον τομέα της ασφάλειας, της οικονομίας, την ε, κοινωνική συμπερίληψη όλων, την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά είναι ουσιώδη για την Ευρώπη. Επίσης πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία της τεχνολογικής αλλαγής για να επιτύχουμε την ευημερία και τη βιωσιμότητα του μέλλοντος για όλους τους συμπολίτες μας. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις, προ τις προκλήσεις ενό ταχαίω μεταβαλλόμενου κόσμου. Πρέπει να δώσουμε και προστασία και ευκαιρίες. Ευαίσθητα θέματα, Όπω το μέλλον του ευρωπαϊκού προπολισμού μετά, ε, μετά το 2020, μπορούν να συζητηθούν μόνο εάν γίνει ευρεία συζήτηση, δημόσια. Αν ακούσουμε προσεκτικά τι ανησυχίε των συμπολιτών μα και αν τι λάβουμε υπόψη μα. Η επικοινωνία πρέπει να ενημερώνει του πολίτε για τη δράση τη Ένωση. Ακόμη και πιο επαναστατικέ ιδέε και λύσει θα αποτύχουν εάν δεν, το, δεν τις αναγνωρίσουν, δεν τις μάθουν όλοι και δεν λάβουν τη στήριξη των συμπολιτών μας. Το πολιτικό όραμα του πλαισίου 21-27 θα είναι σημαντικό για την ανάπτυξή μας σε κάθε επίπεδο, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, για τις επόμενες δεκαετίες. Οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας βρίσκουν σύμφωνος ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τις ε, δαπάνες και με τα έσοδα. Πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση από αυτόν και πρέπει μόλις έχουμε τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περάσουμε σε λεπτομερή συζήτηση. Λοιπόν, να μην πω περισσότερα, να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννους Λεβαντόφσκι και τον κύριο Ζεγάρ που είναι οι συνεισηγητές για τους ίδιους πόρους, για τις παρατηρήσεις τους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είμαστε δύο οι συνεισηγητές αλλά μιλάμε με μια φωνή. Θέλουμε να καλωσορίσουμε τους ε, εθνικούς ε, βουλευτές. Εδώ συζητούμε τα έσοδα τα νέα έσοδα και μάλιστα παρουσία του φίλου Αλέν Λαμασούρ που κάθεται εκεί, τον βλέπετε, και ο οποίος ε, είναι η ζωντανή μνήμη, αν θέλετε, παλιότερων προσπαθειών για τον εξυγχρονισμό και την μεταρρύθμιση της πλευράς των εισόδων του προπολογισμού. Οι απόπειρες αυτές δεν στέφτηκαν πάντοτε με επιτυχία. Αλλά δεν μας αποθάρρυναν αυτές οι αποτυχίες και το ξαναπροσπαθούμε. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε και την Κομισιόν να δείξει τόλμη την προηγούμενη φορά ήμουν εγώ με δύο προτάσεις για το φόρο χρηματοπιστών συναλλαγών και τον απλουστευμένο ΦΠΑ πίσω από τις προτάσεις της Κομισιόν. Υπήρχε και το θέμα της Βρετανικής έκπτωσης όμως τότε και γι' αυτό απάντησαν όχι βρετανικά κατηγορηματικά και έληξε ιστορία εκεί. Υπήρξε λοιπόν ενισχυμένη συνεργασία μόνο για το των πιστοτικών συναλλαγών. Πάντως τώρα το ξαναπροσπαθούμε γιατί ίσως αυτή την ε, περίπτωση το Brexit να μας δώσει ε, ένα περιθώριο, ένα παράθυρο ευκαιριών για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νοπό Προσπαθούμε λοιπόν να και έχουμε και ένα ψήφισμα που θα ψηφίσει αυτήν την εβδομάδα η Επιτροπή Προπολογισμών. Προσπαθούμε να είμαστε τολμηροί αλλά όχι προκλητικοί που σημαίνει ότι δεν προτείνουμε αλλαγή της συνθήκης. Θέλουμε να υπάρχει ε, δημοσιονομική εθνική κυριαρχία γιατί η φορολογική πολιτική είναι προνομία των εθνικών κρατών και εθνικών κοινοβουλίων και έτσι πρέπει να παραμείνει. Ποιο είναι όμως το παράδοξο με το εφιστάμενο σύστημα που είναι και πολύπλοκο και αδιαφανές. Όσο περισσότερη είναι η εθνική συνεισφορά μέσω του εθνικού ακαθάριστου εισοδήματο, τόσο οι χώρε μέλη αυτό το βλέπουν ω κόστο και όχι ω επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό επηρεάζει και τι διαπραγματεύσει. Η καθαρή θέση είναι αυτή που κρίνει την επιτυχία την αποτυχία. Είναι πολύ εύκολο να ασκήσουμε επικρίσεις στο ισχυον σύστημα. Το παράδοξο όμως είναι ότι αυτό το σύστημα που του ασκείται τόση κριτική από τη δεκαετία του 80 παραμένει ιδιαίτερο σταθερό. Βέβαια υπάρχουν και επίμαχα ζητήματα και το πιο επίμαχο θέμα είναι ποιοι είναι, είναι οι υποψήφοι για νέους ίδιους πόρους. Και με τον Ζεράρ Ντεπρέ προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες προτάσεις, ε, δεν είναι και κάποια πρόταση τέλεια. πιστευμένος ΦΠΑ που χωρίς φερτάν στον Πουρσέ ίσως να είναι κάτι πιο εύκολο να περάσει. Φόρος χρηματοπιστών συναλλαγών που δεν είναι ο φόρος Τόμπιν, ούτε καν φόρος χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, αλλά συναλλαγών για να μειωθεί η τάση κερδοσκοπική των χρηματαγορών. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τα νοικοκυριά στις καθημερινές τους συναλλαγές. Επίσης στην πρότασή μας εξετάζουμε και το ενδεχόμενο ε, του εταιρικού φόρου, ένα μερίδιο να μπει ως ίδιος πόρος, ψηφιακός τομέας και για τη χώρα μου το πιο δύσκολο είναι κάτι που θα προωθεί την κλιματική, μάλλον την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Ένας περιβαλλοντικός φόρος δηλαδή. Οπότε στο σχέδιο πρότασής μας, το πιο ουδέτερο που έχουμε προτείνει, είναι ο φόρος προσαρμοσγής ε, στον άνθρωπο που ουσιαστικά αφορά φορολόγηση εισαγωγών από τις χώρες που δεν έχουν ένα σύστημα αντίστοιχο με το δικό μας σύστημα εμπορίας δικαιώματων εκπομπών το ETS. Υπάρχουν και άλλα έσοδα βέβαια που μπορούν να συμπεριληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια είναι προβλέψιμα, συνεισφορές τρίτων χωρών ή φορολόγηση των μισθών των ευρωυπαλλήλων. Αυτά τα έχουμε ήδη και διάφορα άλλα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να ενθαρρύνουμε τον Επίτροπο Έτιγκερ να κάνει προτάσεις για τους ίδιους πόρους. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι. Κύριε Ντεπρέ, εσείς τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως, συμφωνώ με τον συνάδελφο και συνεισηγητή Λεβαντόφσκι. Θα ήθελα να συνοψίσω τη δική μας θέση. Σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, πιο γενικό. Είναι σαφές ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι νέοι πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακούω ορισμένους ε, και εδώ στην αίθουσα ίσως να υπάρχουν τέτοιοι που λένε ότι ο ενωσιακός προπολογισμό είναι ένα πολύ σημαντικό φορτίο που όλο και αυξάνεται. Δείτε τι ε, ποσοστό είναι το αγωνιστικό πρόβλημα σε σχέση με το ΑΕΠ. Το 93-96 ήταν 1,27 ενώ το 2014-2020 σε αυτό το πολιετές ήταν το αντίστοιχο ποσοστό 1,03. Δηλαδή ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σε σχέση με την παραγωγή πλούτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα αυτό. Δεύτερον, ακούω συχνά να γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ των καθαρών εισφορών και των καθαρών δικαιούχων. Έχει και ένα μια δόση αλήθεια σε όλο αυτό, όμως οι καθαροί εισφορείς δεν ε, υπολογίζουν πάντα το τι αυτοί αποκομίζουν από το σύνολο του συστήματος για κάποιες οικονομίες και για κάποιες χώρες. Επειδή έχουμε αυτή την τεράστια νέα αγορά με εναρμονισμένα πρότυπα και κανόνες για προϊόντα και ε, και τη χρήση του κοινού νομίσματος, ε, αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε μηχανική διάκριση μεταξύ των καθών και των καθαρών δικαιωμάτων. Αυτό είναι τεχνητό. Και είναι και λάθος σε ένα βαθμό. Τρίτον, γιατί μιλάμε τώρα για νέους ίδιους γιατί πρέπει να αναπληρώσουμε τις τρύπες, να κλείσουμε τις τρύπες που δημιουργεί το Brexit, και για να καλύψουμε τις νέες προτεραιότητες. Ορισμένοι εξημών μιλήσατε και νομίζω ότι είναι μια κοινή ανησυχία στους περισσότερους από εμάς για την ανάγκη να τα καταφέρουμε καλύτερα σε κάποιους τομείς, όπως για παράδειγμα στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση διαχείριση μεταναστευτικών ροών, αλλά και πολιτική, εσωτερική πολιτική ισορροπία, αν μπορώ να το πω έτσι, για τις εθνικές κοινωνίες. Η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο έγγραφο. Πώς θα κάνουμε πιο αποτελεσματικά τα εθνικά τέσσερα σενάρια, μινιμαλιστικό, τέσσερα δις επτά χρόνια και ένα μαξιμαλιστικό σενάριο μια πραγματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, θα είναι αποτελεσματικός και θα τον διαχειριζόμαστε από εκείνο. 150 δις από τα χρόνια. Αυτές είναι προτάσεις Κομισιόν. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να αποφασίσουμε με βάση τις προτεραιότητες που εμείς θα επιλέξουμε ποια θα είναι τα πρόσθετα μέσα τα οποία θα χρειαστούμε για τα επόμενα χρόνια. Παντού και σε μια ερώτηση, μια απορία. Θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι. Αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν θα πει ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό φόρο που θα τον αποφασίσει. Το είπε και ο Γιάννους. Γιατί η εθνική κυριαρχία είναι κάτι που δεν πρόκειται να ακουμπήσουμε. Θέλουμε να ωφεληθούμε από φόρους και έσοδα που ήδη υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, ΦΠΑ ελπίζουμε ένα αρμονισμένο ΦΠΑ. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ΦΠΑ δηλαδή. Απλά παίρνουμε ένα μερίδιο, ένα ποσοστό που θα το ορίσουμε από κοινού. Και θα το, χρηματο... θα το χρησιμοποιήσουμε για τη χρηματοδότηση του ενωσιακού προπολογισμού. Το ίδιο για την κοινωνοποιημένη βάση φορολόγηση εταιριών. Το ίδιο αν συμφωνήσουμε αύριο για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το ίδιο αν συμφωνήσουμε για κάποιου πράσινου φόρου, οικολογικού φόρου. Δεν θα δημιουργήσουμε λοιπόν ευρωπαϊκού φόρου ένα ευρωπαϊκό φορολογικό επίπεδο, αλλά θα αξιοποιήσουμε φόρους που ήδη υπάρχουν ε, σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, για όσους ανησυχούν, γιατί κάποια κοινοβούλια και κάποιοι συνάδελφοι ξέρω ότι πιστεύουν ότι πιο δίκαιη συνεισφορά είναι εθνική, συνεισφορά που υπολογίζεται με βάση το εθνικό ακαθάριστο εισόδημα. Δεν θα καταργηθούν οι εθνικές εισφορές, απλά θα μειωθεί σχετική τους ε, αναλογία στο ενωσιακό προπολογισμό. Και ιδανικά θα θέλαμε σε αυτή την επταετία να μειωθούν οι εθνικές εισφορές κατά 40% και τη σκητάλη να την πάρουν νέοι ήδη πόροι για τους οποίους μίλησε ο Γιάννους και που όλο αυτό θα είναι ένα ισορροπημένο πακέτο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά είχα εγώ να πω στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντεπχέ. Ο κύριος Αλάν Λαμασούγ έχει τώρα το λόγο, ε, μέλος της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να σταθώ σε ορισμένα σημεία τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί από τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή, ε, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση αυτού του ενωσοκοπού προπολογισμού, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε πλέον να αποφύγουμε γιατί υπάρχει ένα ψαλίδισμα μεταξύ των ε, συνηθισμένων εσόδων που θα πέσουν ε, θεαματικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και από την άλλη την αύξηση των αναγκών. Έχουμε ήδη μια αύξηση των ευρωπαϊκών ευθυνών και αρμοδιοτήτων που έχει ήδη αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Συμβούλιο, από τα κράτη-μέλη και έχει κυρωθεί από τα κοινοβούλια και το εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, την καταπολέμηση της θερμοκρατίας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη νέα εταιρική σχέση που θα πρέπει να αναπληρώσουμε με την Αφρική. Για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που είχαμε να κάνουμε μέχρι τώρα, έχουμε ε, δημιουργήσει ένα ταμείο με συγκεκριμένε ε, μεταβλητέ για κάθε νέο πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσουμε όμω αυτό το ε, σπάταλο σύστημα και να αναθεωρήσουμε τον κοινό μας χρηματοδοτικό μηχανισμό. Αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι και καμία επανάσταση, όπως ανέφερε ο κύριος Δεπχέ. Η... η βασική ευθύνη και κυριαρχία, η οικονομική κυριαρχία παραμένει στο εθνικό επίπεδο, δεν πρέπει να μεταφερθεί στο ευρωπαϊκό, όμως εξετάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, μία ε, συλλογικότητα επικρατιών, όπως στη Γαλλία, στη χώρα μου, ε, δίνουμε το δικαίωμα στις περιφέρειες και στις πόλεις να έχουν ιδίους πόρους και πάλι όμως εθνική είναι η κυριαρχία στο οικονομικό επίπεδο, εξετάζεται και ελέγχεται από το Κοινοβούλιο. Ε, απλώς αφήνει τη δυνατότητα στις πόλεις και στις περιφέρειες να επιβάλλουν ορισμένους ε, φόρους με συγκεκριμένα ποσοστά που έχουν προκαθοριστεί αυτός είναι ο μηχανισμός. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κατά τη διάρκεια των 21 ετών της ΕΟΚ τότε, η ευρωπαϊκή κοινότητα λοιπόν λειτουργούσε αποκλειστικά και μόνο επί αυτή τη βάση των ε, ιδιών πόρων και χωρίς εθνική εισφορά. Είχαμε τότε λοιπόν τους ίδιους πόρους, ε, τους δασμούς, τότε που ήταν ακόμα προστατευτική η προσέγγιση. υπήρχε ακόμα και φόρος που τώρα θα χαρακτηρίζαμε ως ε, ομοσπονδιακός, ε, που ε, τον δεχόντουσαν όμως όλοι και αφορούσε έναν φόρο που είχε προκύψει από τη συνθήκη για τον άνθρακα και το χάλεβα και λειτουργήσε αυτό το σύστημα για 20 χρόνια. Στην πορεία εξελίχθηκε βέβαια εφόσον τώρα έχουμε χρηματοδότηση από τις εθνικές συνεισφορές. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι επαναστατικό, επιστρέφουμε σε αυτά που κάναμε στο παρελθόν. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας λοιπόν. Συμμερίζομαι τώρα τις προτάσεις ε, των εισηγητών. Ήθελα μόνο να επισημάνω ότι όπως και να έχει, εάν έχουμε την ομοφωνία των κυβερνήσεων και των Υπουργείων Οικονομικών για τους επιμέρους πόρους, τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν τον τελευταίο λόγο και το καθένα από αυτά θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει δικαίωμα ανησυχηρίας. Οπότε αυτό πρέπει να σας καθεσυχάσει. Μια τρίτη παρατήρηση. Πολύ σωστά το ανέφερε και ο πρόεδρος Αχτσουή προηγουμένως. Πρέπει να φροντίσουμε για κάθε ευρώ, επιπλέον ευρώ που δαπανάτε στις Βρυξέλλες, να υπάρχει τουλάχιστον ένα ευρώ εξοικονόμησης στην εθνική οικονομία. Και αν ε, αποφασίσουμε ότι η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται αποκλειστικά ή περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μεταφέρουμε και τα αντίστοιχα, ε, τους αντίστοιχους πόρους μέσω φορολογικών πόρων. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στον φορολογούμενο, γιατί σε τελική ανάλυση ο φορολογούμενος είναι αυτός που καταβάλει τους φόρους και έτσι καλύπτονται οι πόροι ε, για την ε, εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Οπότε δεν θα πρέπει τελικά να αυξηθεί ε, το φορολογικό άχθος. Αντιθέτως, θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά μας. Γι' αυτό προτείνω ε, και τα εθνικά ελεγκτικά μας συστήματα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ε, διασφαλίζουν, να επαληθεύουν ότι κάθε φορά που μεταφέρεται μία εθνική αρμοδιότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή η αρχή της επικουρικότητας θα τηρείτε και θα επαληθεύεται για κάθε ευρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που τηρήσατε και το χρονικό όριο. Να περάσουμε τώρα στους προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο Σλάχτε, από την Πολωνία. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ακούσαμε προηγουμένως ε, ότι τα εθνικά κοινοβούλια ε, μπορούν να μιλάνε ελεύθερα. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να σας ε, δώσω την άποψη της πολωνικής κυβέρνησης του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Είμαστε έτοιμοι για να συζητήσουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και γνωρίζουμε τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν μιλάμε μόνο για τη στρατιωτική ασφάλεια, μιλάμε και για την ενεργειακή ασφάλεια, επί παραδείγματι. Και πραγματικά η θέση μας σε ό,τι αφορά τον δεύτερο North Stream αγωγό είναι πολύ ξεκάθαρη. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή των προτεραιοτήτων θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τους στόχους ε, μεταξύ άλλων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη προσέγγιση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περικοπεί ο νοσιακός προϋπολογισμός. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι προτάσεις του Επιτρόπου Έτιγκερ. Που προτείνει ποσοστό 1,1 σε σχέση με το ΑΕΠ για τον ενωσιακό προπολογισμό. Σε ό,τι διαφορά τους ίδιους πόρους, πιστεύουμε ότι πρέπει να αυξηθούν. Σε αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιόν Βίσελ από τη Σουηδία. Den svenska positionen är känd. Λοιπόν, στηρίζουμε σταθερά την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να σας πω ότι η στήριξη του ευρωπαϊκού, συγγνώμη, του σουδικού λαού έχει αυξηθεί μετά το Brexit. Όμως δεν μπορούμε τόσο εύκολα να πείσουμε το σουδικό λαό να αυξήσει την συμβολή του στον ενωσιακό προπολογισμό. Εδώ θα υπάρξει αντίσταση. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που θα πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω. Αλλά η, το Brexit πρέπει να οδηγήσει στο να ε, μειωθεί η χρηματοδότηση της Ένωσης. Δηλαδή, για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή ή την ε, προσφυγική κρίση, πρέπει να κινητοποιηθούν εθνικοί πόροι. Στην ε, γεωργική πολιτική επίσης θα μπορούσαν να υπάρξουν εξοικονομήσεις. Και αν θέλουμε να αυξηθούν οι ε, φόροι, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως ε, θα υπάρξει ανάκαμψη και περισσότερη κοινωνική Ευρώπη. Να αναλογιστούμε εάν η αύξηση των ενωσιακών ε, πόρων θα σημάνει μείωση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα χωρίς να περιορίσουμε την, ε, χωρίς να περιορίσουμε τους, ενωσιακούς, τους εθνικούς φορολογικούς πόρους. Χωσέφ Μανώλη Φερνάνδες από την Πορτογαλία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Και πολύ εύκολα μπορεί να γλιστρήσει προς τον λαϊκισμό. Ορισμένοι θέλουν ναι μεν να αυξηθεί ο νοσιακός προϋπολογισμός αλλά μετά λένε όχι δεν θέλουμε νέους ίδιους πόρους. Άρα θα χρειαστούν μεγαλύτερες εθνικές συνεισφορές. Άρα περισσότερη φορολογία των πολιτών της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να αυξηθεί ο ενωσιακός προπολογισμό, ο πιο λογικός τρόπος για να το κάνουμε είναι, είναι να βρεθούν πόροι που δεν θα επιβαρύνουν τους πολίτες. Ορισμένοι άλλοι θέλουν να διατηρηθεί το υπάρχον σύστημα, δηλαδή οι εθνικές συνεισφορές. Όπου οι Υπουργοί Οικονομικών θεωρούν ότι είναι ιδιοκτήτες του ενωσιακού προπολογισμού. Και ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι τους ανήκει περισσότερο από τους άλλους, από ότι ανήκει στους άλλους. Αλλά δεν είναι σωστέ αυτέ οι διακρίσει, γιατί έτσι κάνουν διάκριση μεταξύ καθαρών συνεισφορέων και καθαρών ε, ωφελουμένων. Αλλά επενθυμίζω, το 85% ε, του προπολογισμού ε, προέρχεται από τα κράτη-μέλη. Η Γερμανία και η Γαλλία πληρώνουν 38% του προπολογισμού των 28. Όμως ε, ο προπολογισμό δεν είναι ιδιοκτησία των Υπουργών, αλλά όλων των πολιτών και όλα τα κράτη-μέλη υποφελούνται από τις δαπάνες του. Ακόμη και όσοι είναι καθαροί συνεισφορείς, ωφελούνται από άλλα δημόσια αγαθά που έχουμε. Δεν ξέρω αν ε, γνωρίζει ο πολίτης ότι το 94% του προπολογισμού είναι επενδύσεις που επιστρέφουν κατά 80% στα κράτη-μέλη. Κάποτε λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και το κόστος της κατάργησης των πολιτικών που έχουμε. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι καθαρός συνεισφορέας, κατάλαβε πολύ καλά πόσο θα του κοστίσει η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. θα του κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι του κοστίζει τώρα η συμμετοχή του. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Η κυρία Σαμπίν Τιλάι. Σας παρακαλώ δύο λεπτά να μην υπερβαίνετε το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθώντας αυτή τη συζήτηση διαπιστώνω ότι υπάρχει πρόβλημα πολιτικής βούλησης. Ε, γενικόλογα όλοι λέμε βεβαίως πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Αλλά τώρα θεωρούμε ότι έχουμε κοινό πεπρωμένο ως ένωση. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν και οι φορολογούμενοι. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Δεν μπορούμε πλέον να το αποφύγουμε. Κοιτάξτε, εμεί ω Εθνικό Κοινοβούλιο, όταν αποφασίζουμε τον προπολογισμό, είμαστε υπόλογοι στους ε, πολίτες μας. Η Γαλλία πρότεινε ε, μια διαδικασία διαβούλευσης των πολιτών. Ο πρόεδρος Μακρόν το πρότεινε. Το αποδέχθηκαν 25 κράτη-μέλη. Γιατί να μην θέσουμε και εμείς αυτό το θέμα να ρωτήσουμε τους ε, συμπολίτε μας ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο και έτσι θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες για να αποφασίσουμε τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζαμπέλ Τομάς, εισηγήτρια για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα λοιπόν θέλω να πω ότι και στο έργο της ομάδας υψηλού επίπεδου ε, στην οποία συμμετείχε ο κ. Ναμασούχα αλλά και συνολικά στο Κοινοβούλιο εργαστήκαμε προκειμένου να βρούμε και να συγκλίνουμε προς ε, έναν στόχο. Θα πρέπει να είναι τα κρατημέλη και το Εθνικό Κοινοβούλιο δικαιούχοι των ίδιων πόρων. Θα πρέπει λοιπόν και να ε, μειώσουν, να ελαφρύνουν το ευρωπαϊκό βάρος των εθνικών προπολογισμών. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί μπορούμε ε, να διευρύνουμε το ε, περιθώριο ευελιξίας των εθνικών προλογισμών και των εθνικών κοινοβουλίων. Δεύτερον, οι προτάσεις του εισηγητή δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη μη επιβολή περαιτέρω επιπρόσθετων βαρών στον Ευρωπαίο Φορολογούμενο θέλουν ε, να αντιμετωπίσουν εκείνους που δεν συμβάλλουν ε, στον δημόσιο καρβανά, επενδύοντας στις υποδομές, στην κατάρτιση και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η άγουσα που προτείνουμε εμείς. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Πολύ σύντομα, αν θέλουν οι ομιλητές να πάρουν πάλι το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Για ορισμένε καταληκτικέ παρατηρήσει. Εντάξει. Μιλούμε για νέους ιδίους πόρους, όμως δεν πρέπει εδώ να μιλήσουμε και τις εθνικές εισφορές. Αυτό είναι το μόνο δίκαιο, γιατί έχει να κάνει με τις ε, πλούσιες και λιγότερο πλούσιες χώρες. Και αυτό είναι κάτι προβλέψιμο με βάση την αυτόματη προσαρμογή. Η ήδη πόρη δεν είναι τόσο προβλέψιμος μηχανισμός και μετά είναι και θέμα πολιτικής βούλησης και έχετε ε, δίκαιο ότι είναι καθοριστική σημασία η πολιτική βούληση. Τώρα, Πώς ε, μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον με την Βουλγαρική Προεδρία, καθώς θα εξετάζουμε την πρόταση του Ettinger, ελπίζω κάτι να γίνει. Είχαμε και την Αυστρία που δεν ήταν ε, πραγματικά υπέρμαχος ε, των ίδιων πόρων, όμως είναι ένα καθοριστική σημασία σε εξάμεινο, αν θέλουμε να οριστικοποιήσουμε αυτό το φάκελο ο ρόλο τη Αυστρία θα είναι πολύ σημαντικό ε, σε ό,τι αφορά το εξάμεινο του 2018 και εδώ τίθεται το ερώτημα. Πώ μπορούμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Ε, oui, Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Από αυτή τη σύντομη ανταλλαγή απόψεων νομίζω ότι προέκυψε το εξή συμπέρασμα. Για να αιτιολογήσουμε τους πόρους ε, που ζητούμε και τις δαπάνες που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει αρχικά να συμφωνούμε ε, να συμφωνήσουμε επί των κοινών μας ε, στόχων. Τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε από κοινού. Και μέσω αυτής της σύντομης συνταλλαγής απόψεων και κατά το παρελθόν αλλά και σήμερα βλέπουμε ποια θα είναι οι, μεγα... ποιες θα είναι οι μεγάλες προκλήσεις για να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για το επόμενο ΠΔΠ. Πώς θα τα καταφέρουμε και εμείς και τα κράτη-μέλη να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των πολιτικών που θέλουμε να εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε, τη συνοχή της γεωργικής πολιτικής και από την άλλη να αντιμετωπίσουμε και τις νέες προκλήσεις που θα ζητούν όλα και περισσότερους πόρους και συνεργασία αν θέλουμε να καλύψουμε και να πραγματοποιήσουμε όλους τους στόχους μας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντεπχέ. Ζητώ συγγνώμη τον κύριο Λαμασούχ. Ε, υπενθυμίζω σε όλους και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι το σλόγγαν μας, το μότο μας είναι η ισχύς εν τη ενώση. Αν όλοι λοιπόν ε, ε, λειτουργούμε και παρότι όλοι λειτουργούμε σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο πρέπει να ενεργούμε από κοινού. Υπενθυμίζω ότι το δείπνο είναι στις 7 το απόγευμα στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σε πέντε λεπτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαχτσί, περιμένουμε πολλά από την Βουλγαρική Προεδρία.